Οι αρμόδιες αρχές ε, της ε, Γαλλικής Δημοκρατίας μου ζήτησαν ε, άρση της ασυλίας των κυρίων Στίβ Μπρουά και της κυρίας Σοφή Μοντέλ στα πλαίσια μιας έρευνας που ξεκίνησε από το δικαστήριο της Ναντέρ. Βάσει του κανονισμού τα αιτήματα αυτά έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Θυμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου